Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Λυπάμαι που περιμένατε. Έπρεπε να τελειώσουμε με τη συνάντηση των ε, συντονιστών. Θα πάμε αμέσως προς την ημερήσια διάταξη, δηλαδή την ψηφοφορία. Ως προς την ε, βιοπικιλότητα και τα οικοσυστήματα, τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων για την ανάπτυξη των στόχων της χιλιετίας. Ψήφισμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Α, ομοφωνία. Ωραία. Αποχές. Καμία. Άρα εγκρίνεται ομοφόνος. Ωραία. Τώρα θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι στο Στρασβούργο στις 5 Οκτωβρίου θα έχουμε μία συνοπτική, ένα συνοπτικό ψήφισμα, ένα συγκεφαλαιωτικό ψήφισμα και στις 13 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Η επόμενη ψηφοφορία αφορά την Συμφωνία Αλίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νήσων του Σολομώντα. Υπάρχουν δύο τροπολογίες από τον κύριο Αρσένη που δεν είναι παρόν. Τροπολογία παριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ομόφωνα επίσης. Τώρα ψηφίζουμε την γνωμοδότηση όπως έχει τροπολογηθεί υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ομόφωνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Then we Στη συνέχεια Έχουμε την γνωμοδότηση Μπέρμαν για τον χρηματοοικονομικό κανονισμό. Χτες η Επιτροπή δεν μπόρεσε να γνωμοδοτήσει. Γι' αυτό αποφασίσαμε να τους ε, χορηγήσουμε αυτό το χρόνο, αυτό το διάστημα. Ο κύριος Μπρένταν Κόγκαν από την Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού είναι εδώ. Θα ήθελα να σχολιάσει την γνωμοδότηση Μπέρμαν. Καλημέρα σας. Είπε ότι θα είναι στις 10 και 20 και δεν είναι ακόμα 10 και 20. Μπορείτε να περιμένετε 5 λεπτά. Εντάξει, θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο στο μεταξύ. Άρα ας δούμε τον δημοκρατικό έλεγχο μέσα στα πλαίσια του γενικότερου ε, προγραμματισμού. Πρόκειται για την ε, ομάδα εργασίας Α μέσα στα πλαίσια της Επιτροπολογίας, η Επιτροπή ΔΕΒΕ ελέγχει τις δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στα πλαίσια του Μέσου Ανάπτυξης και Συνεργασίας. Η Ομάδα Εργασίας Α έχει αποτιμήσει το στρατηγικό έγγραφο για την Ινδονησία και τα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Κεντρικής Ασίας. Ο κύριος Νιούσερ είναι πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Α και του δίνω το λόγο για έξι λεπτά. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεδρίασε η ομάδα Α με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι 24 Ιουνίου για να συζητήσει το έγγραφο της ενδιάμεση αναθεωρή σχετικά με το έγγραφο στρατηγική και τι δραστηριότητες ε, εκπαίδευσης για το 2010 στην Κεντρική Ασία στα πλαίσια του προγράμματος δράσης. Ε, υπήρχαν και μέλη της Ασιατικής Αντιπροσωπείας στη συνεδρίαση. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Ε, υπήρχαν μέλη των αντιπροσωπιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνεδρίασή μας και μας ενθάρρυναν δράτω με τις ευκαιρίες για να καλέσω όλα τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά της ομάδας εργασίας, για να αφιερώσουν λίγο από το χρόνο τους σε ένα από τα βασικά καθήκοντα κατ' εμέ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή άσκηση δημοκρατικού ελέγχου σχετικά με την απόφαση που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η άσκηση αυτού του δικαιώματο μα δίνει την ευκαιρία να δούμε πώ εφαρμόζονται στην πράξη τα νομοθετήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι με καλύτερο τρόπο μπορούμε να ε, προαγάγουμε τι πολιτικέ προτεραιότητε του Κοινοβουλίου. Στα πλαίσια του εγγράφου στρατηγική για την Ινδονησία, ε, θα έλεγα ότι το πρώτο τμήμα το έχουμε αναλύσει ήδη στην Επιτροπή Ανάπτυξης το 2007 και έκτοτε αντιλαμβανόμαστε ότι σημειώθηκε η ικανοποιητική πρόοδος ως προς την υλοποίηση ε, της Συμφωνίας Συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδονησία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει δεόντως υπόψη τις προηγούμενες παρατηρήσεις που έγιναν το 2007 στο Κοινοβούλιο και έτσι υπάρχει ένα ειδικό τμήμα για παρέμβαση στον τομέα των κλιματικών αλλαγών και άλλες δραστηριότητες ε, ε, για να ε, προωθήσουμε τις εθελοντικές συμφωνίες, δηλαδή ενισχυμένη διακυβέρνηση και ενισχυμένες εμπορικές συναλλαγές. Ένα από τα εκρεμή ζητήματα στην Ινδονησία είναι το θέμα του AIDS και η βασική ιατριοφαρμακευτική περίθαλψη. Βάσει της ομάδας εργασίας Α θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα μέσα στο έγγραφο στρατηγικής σε αυτούς τους τομείς. Επίσης, ε, διαπιστώνουμε ότι ο τομέας της υγείας ε, δεν είναι βασική προτεραιότητα για το έγγραφο στρατηγικής που καλύπτει την περίοδο 2007-2013. Ε, παρέχεται βοήθεια μέσω του Παγκοσμίου Ταμείου για το AIDS προς την Ινδονησία καθώς και για την Ελλονοσία. Συγκεκριμένα η Ινδονησία είναι η δεύτερη σε μέγεθος χώρα, ο δεύτερος αποδέκτης κονδυλίων 308 εκατομμύρια στο σύνολο ε, εκ των οποίων τα 97 είναι για την καταπολέμηση του AIDS και καλύπτονται 12 περιφέρειες από τις 43 ε, για την προληπτική δράση, την περίθαλψη, την υποστήριξη και τις θεραπευτικές αγωγές μέχρι το 2014. Η ομάδα εργασίας επίσης σημείωσε ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς παραμένει πρόκληση στην Ινδονησία και Γι' αυτό καλούμε την Επιτροπή Ανάπτυξης να συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα της διαφάνειας και λογοδοσίας. Ε, επ' αυτού είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή, να υπενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λαμβάνει τακτικά τις εκθέσεις σχετικά με τη δημοσιονομική στήριξη ε, της ρήτρης διασφάλισης και την αιρεσιμότητα. Λοιπόν, τα πορίσματα και οι συστάσεις μας προς την Επιτροπή ανάπτυξη. σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας διαβούλευσης συμπεριλαμβάνονται μέσα στο έγγραφο και η ομάδα εργασίας Α συστήνει προς την ε, Επιτροπή ανάπτυξη ε, να ε, λάβει γνώση του εγγράφου στρατηγικής για την Ινδονησία και σας καλούμε να αποδώσετε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στις επόμενες εκθέσεις όπου θα δείτε την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί στον τομέα της υγείας ε, σε σχέση με τους στόχους της χιλιετίας. Επίσης, ε, καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης ε, να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη αυτή την ανάγκη του Κοινοβουλίου, δηλαδή να λαμβάνει το Κοινοβούλιο τακτικές εκθέσεις σχετικά με την αιρεσιμότητα και την πρόοδο που σημειώνεται, ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής δημοκρατικός έλεγχος για την εφαρμογή του εγγράφου στρατηγικής μέσα από τα ετήσια προγράμματα δράσης. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Θα ήθελε κάποιος ε, συνάδελφος να σχολιάσει αυτές τις συστάσεις της ομάδας εργασίας Α για την εκπαίδευση, για το AIDS, για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν σε σχέση με την Ινδονησία. Συμφωνείτε λοιπόν με τα συμπεράσματα που μας προτείνει η ομάδα εργασίας Α. Ναι, δεν υπάρχουν ενστάσεις πάρα πολύ ωραία, οπότε θεωρώ ότι εγκρίθηκαν τα συμπεράσματα και κλείνει και η προθεσμία για το δικαίωμα ελέγχου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, εργαστήκατε με εξαιρετικό τρόπο. Τώρα... Για τρίτη φορά στρέφομαι ε, προς τον συνάδελφό μου, τον κύριο Μπέρμανε, για τον δημοσιονομικό κανονισμό και με χαρά θα υποδεχτούμε τον κύριο Κόγκμαν από την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ προϋπολογισμού που θα αποφανθεί για την έκδοση του κυρίου Μπέρμαν. Α, ο κύριος Νάζης ξαναζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Part, Νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να παρουσιάσω το δεύτερο μέρος ε, για την ομάδα εργασίας Α σχετικά με το πρόγραμμα Έρασμος. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόγραμμα Erasmus που ε, προτείνεται για την κεντρική ε, Ασία που συνάδουν με το πρόγραμμα 2007-2010 και τους στόχους της ε, DCI καθώς και τις προτεραιότητες. Η ομάδα εργασίας παρακαλεί την ε, Επιτροπή ε, να εξετάσει τις διάφορες δραστηριότητες διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διευκρινίσει ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα είναι τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα των κρατών μελών που χρηματοδοτούνται για τις δημοσιεύσεις και για τα γενικά έξοδα και επιπλέον τα κράτη αυτά είναι, ε, έχουν τους μόνους οργανισμούς που μπορούν ε, να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Tempus. Θα πρέπει να σας πω ότι ε, θα θέλαμε να καλύψουμε τους διάφορους οργανισμούς κατά τρόπον ώστε ε, να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους ε, στόχους και ε, να συνδυάσουμε ε, ε, τους στόχους αυτούς με τη συνεργασία των κρατών μελών ε, και την ανταλλαγή αρμοδιοτήτων διότι δεν πρέπει η χρηματοδότηση αυτή να, χρηματο... να χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, έχουμε εξετάσει ε, την ε, κινητικότητα του προγραμματος ερεσμους Έρασμους 2008-2010 που δεν χρηματοδοτείται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 100% της συμμετοχής είναι από τρίτες χώρες. Τα συμπεράσματά μας είναι ότι τα μέτρα τα οποία προτείνονται πρέπει να τύχουν στηρίξεως αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης την κατάσταση στην ε, Νότια Ασία ιδίως όσον αφορά το Ταζικιστάν και τις ε, χώρες όπου πρέπει να αυξηθεί η δραστηριότητα, η Επιτροπή Ανάπτυξης σε αυτό το σημείο βάσει των στοιχείων που έχει και των απαντήσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως οδηγεί την ε, ομάδα εργασίας να προτείνει να μην υπάρχει ε, περιορισμός της δράσεως του πρόγραμμα Έρασμος το 2010 και να εφαρμοστεί το άρθρο 35. Ζητείτε επίσης να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να εξασκήσουν το δικαίωμα εξετάσεως και η Επιτροπή να παρουσιάσει μία επισκόπηση των μέτρων που προβλέπονται στην Κεντρική Ασία. Ευχαριστώ. Τώρα θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή αν συμφωνεί με τις, τα συμπεράσματα της ομάδος εργασίας και ε, θεωρώ ότι έχει λήξει ε, η προθεσμία για την εξέταση. Και επανέρχομαι για τέταρτη φορά στην ε, γνωμοδότηση του κυρίου Μπέρμαν αντιλαμβάνουμε ότι ο κύριος Κριστόφερσεν, σύμβουλος της Βαρόνης Άστον, είναι επίση στην αίθουσα και ελπίζω ότι μετά από το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Βέρμαν θα λάβει τον λόγο. Μάλλον πριν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, η Επιτροπή εξέτασε τις διάφορες κοπιές και όπως είπατε λέγομαι ε, Μπρένταν Κούγκαν, είμαι εθνικός εμπειρογνώμονας ε, που εργάζεται με την Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και εξετάζοντας τις προτάσεις και την γνωμοδότηση του κυρίου Μπέρμαν καθώς επίσης και τα θέματα τα οποία θίγει που λαμβάνουν υπόψη την αιτιολόγηση στην παράγραφο 3 ε, μας βρίσκουν απολύτως ε, σύμφωνους διότι θεωρούμε ότι η ακεραιότητα θα εμπεδοθεί εις την υπηρεσία και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση. Όσον αφορά την πρόταση, πολλά από τα θέματα αυτά μου φαίνονται πολύ λογικά και βελτιώνουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για αυτό και μπορούν να αναπτύξουν ορισμένα σημεία της πρότασης τουλάχιστον εγώ έτσι αξιολογώ τις ε, προτάσεις ε, του κυρίου Μπέρμαν. Θα είμαι όμως λίγο πιο προσεκτικός σχετικά με την ε, δεύτερη τροπολογία διότι ε, με συγχωρείτε ουσιαστικά ξεκινώ από το άρθρο 12 όπου πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη τα θέματα αυτά. Ένα από τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι όπου ε, αναφερόμαστε εις ε, τα λειτουργικά έξοδα και γι' αυτό ουσιαστικά ε, προτείνουμε εδώ σχετικά με τα αποθέματα να υπάρξουν συζητήσεις με τους συναδέλφους αλλά ουσιαστικά αυτές είναι, αυτά είναι τα σχόλιά μου σχετικά με την πρόταση θεωρώ ότι είναι πολύ καλή Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χαιρετίζει και εκφράζει μόνο αυτή την επιφύλεξη σχετικά με τη δεύτερη τροπολογία. Κύριε Μπέρμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για το σχόλιο αυτό. Θα ήθελα να κάνω μια επιπλέον ερώτηση. Ε, έχετε υπόψη σας ότι η διατύπωση ε, στην ε, παράγραφο 2 είναι ταυτόσιμη με αυτήν της κυρίας Γκρέσλε στην Επιτροπή Προπολογισμού. Εκφράσατε και εκεί την ίδια επιφύλαξη. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα μέχρι σήμερα το πρωί σε 9 η ώρα ότι εγώ θα παριστάμουν εδώ. Οπότε θα επανέλθω σε εσάς για αυτό το θέμα. Μην ανησυχείτε έρχεται, λέει ο είναι κάτι το οποίο έχω συναντήσει επανειλημμένος. Κύριε Χριστόφερσεν, χαίρομαι ιδιαίτερος που είσαστε εδώ και είναι πολύ σημαντικό, σημαντική η παρουσία σας εδώ, οπότε σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω τώρα λοιπόν να σας δώσω το λόγο για να σχολιάσετε τη γνωμοδότησή μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι εδώ και λυπούμε που έχουν υπάρξει ορισμένες παρανοήσεις σχετικά με την παρουσία μου, διότι αυτή τη στιγμή ε, δύο άτομα ασχολούνται με την κατάρτιση της υπηρεσίας αυτής, γι' αυτό και δεν μπορούμε συγχρόνως να είμαστε παντού όπου θα έπρεπε να είμαστε. Η Επιτροπή όμως αυτή είναι πολύ σημαντική για την κατάρτιση της EAS. Στη συνέχεια θα είμαι πάρα πολύ σύντομος ε, αλλά ε, από την αρχή η ύπατος ε, εκπρόσωπος ήθελε να εξασφαλίσει ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν πρέπει να μειώσει τη δημοσιονομική πτυχή της εξωτερικής δράσης της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Και πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με το βασικό κανονισμό είχαμε λάβει πολλές προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συνέβαλαν εις την διατύπωση του κανονισμού που, επί του οποίου γνωμοδοτεί τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που αναφέρεται και σε άλλα θέματα πέραν του δημοσιονομικού ελέγχου. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι σήμερα οι ενέργειες ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση και δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό το θέμα. Έχω όμως περισσότερο μία ερώτηση από τη μία αντίθεση σχετικά με το ότι προτείνεται στην ε, δεύτερη τροπολογία διότι αν μιλάμε για λειτουργικά έξοδα είναι λογικό η Επιτροπή και ο, ο, ο οικονομικός ελεγκτής να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει ε, τα στοιχεία αυτά εντός και εκτός της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Ε, οπότε ε, εάν υιοθετήσουμε την τροπολογία η κατάσταση αλλάζει ε, και σύμφωνα με το συμβιβασμό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι υπεύθυνη για τις διοικητικές της πράξεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα έχουμε κάποια επαλήθευση της δεύτερης τροπολογίας γιατί αναφέρεται το όνομά μου ε, και δεν ξέρω εάν θα διατηρηθεί ή θα διαγραφεί. Μπρένταν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εντός ε, λεπτών όταν θα φύγω από το, την αίθουσα αυτή θα το εξετάσω. Άλλοι συνάδελφοι. I would uh, like to say thank you very much. Τότε σας ευχαριστώ για όλες σας αυτές τις ενέργειες και ε, θα παρακολουθούμε και θα επαγρυπνούμε ε, για το ε, τομέα σας και προσβλέπουμε στην παρουσία της Βαρόνης Άστον συχνά στην Επιτροπή μας για να μας ενημερώνει για το τι κάνει. Και θα θέλαμε βέβαια και κάτι παραπάνω, αλλά ε, τουλάχιστον αυτό θα μείνει στα πλαίσια του διαλόγου μεταξύ της υπηρεσίας εξωτερικής ε, ενεργείας και ε, ημών. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς έχει η πραγματικότητα. Η Βαρόνη Άστον πρέπει να μεταβεί από μία επιτροπή σε τουλάχιστον τρεις άλλες Δηλαδή, αντί για εκπρόσωπος της ΚΕΠΑ, θα γίνει, αντί εξωτερική εκπρόσωπος, θα γίνει εσωτερική εκπρόσωπος ως προς τις εργασίες της ΕΙΕΒ. Αναγνωρίζω ότι θέλουμε να ε, δούμε, να βλέπουμε συχνά τη Βαρόνη, είναι εξαιρετική στην εργασία της, αλλά έχει και εξωτερικές ευθύνες και όταν τις επιτρέπουν οι εξωτερικές υποχρεώσεις θα επισκέπτεται τις επιτροπές. Αλλά η εύκολη επιλογή είναι να καθόμαστε και να επικρίνουμε. Και... και θα πρέπει λοιπόν να χαλαρώσουμε, να απολαύσουμε το καλοκαίρι πριν προβάλλουμε άλλες απαιτήσει ε, προς τη Βαρόνη. Άρα είσαστε πολύ πιστός φίλος της, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο θέμα είναι η ανθρωπιστική βοήθεια και η ανοικοδόμηση της ΑΙΤΙΣ. Τι έχει να μας πει η Επιτροπή που επισκέφθηκε την ΑΙΤ. Ο κύριος Στίφλερ, μάλλον η, η Μισελ Στίφλερ ήταν ε, εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας έξι μήνες μετά από, την, ε, από το σεισμό η ΑΕΤ αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Ε, κυρία Στίφλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι Πράγματι μεταβήκαμε στην ΑΙΤΗ στα τέλη Ιουνίου μέσα στα πλαίσια των εργασιών ΔΕΒΕ ε, ε, με τους κυρίους ε, Ρινάλντι και Τιρολιά για να δούμε πώς έχει η διαδικασία ανοικοδόμησης και η χρήση των μέσων μετά από την το σημό τη 12 η Ιανουαρίου. Ευχαριστώ την κυρία Κρυσταλίνα Τζόρτζεβα, την Επίτροπο και την αντιπροσωπεία της, την αντιπροσωπεία μας στο Πόρο Πρένς που εργάζεται κάτω από δυσχερείς συνθήκες και επιτύχαμε στις εργασίες μας. Μας απασχολεί το θέμα των πόρων της αντιπροσωπείας τη στιγμή που όλοι οι φορείς ανοικοδόμησης διπλασιάζουν ή τριπλασιάζουν το προσωπικό. Χρειάζεται ενίσχυση των πόρων για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση τον, του σεισμού. Έξι μήνες μετά τον σεισμό η κατάσταση είναι ανησυχητική. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση κατεπίγουσας ανάγκης. Δυστυχώς η ζωή δεν μπορεί να ξαναρχίσει και υπάρχουν ε, χιλιάδες ε, ε, τόνοι χαλασμάτων. Οι μη κυβερνητικέ δρούν και έτσι συνειδητοποιήσαμε το εύρος της καταστροφής. Μεταβήκαμε σε πολλές αστικές περιοχές που είναι τεράστιοι καταβλισμοί με εκατοντάδες ανθρώπους. Μία δεύτερη μέρα αφορούσε την κατάρτιση και την προστασία του παιδιού με ένα πρόγραμμα στη Μύρμπαλέ που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα τραφή. Πάρα πολλά σχολεία καταστράφηκαν, γύρω στα 4.900 σχολεία καταστράφηκαν και έπρεπε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της χώρας οι ανθρωπιστικές προκλήσεις είναι τεράστιες. Χρειάστηκε 1,5 ε, δις ε, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και 1.200 σημεία καταβλισμών εγκρίθηκαν στην πρωτεύουσα. Έπρεπε να ανταποκριθούμε με το σύστημα των clusters. Αυτό το σύστημα όμως έδειξε τα όρια του. Εξαιτία των προκλήσεων, των ανθρωπιστικών προκλήσεων, επειδή υπάρχει ε, μεγάλη πυκνότητα στα αστικά κέντρα θα έπρεπε ο απολογισμός να λάβει υπόψη και τα μη ορατά αποτελέσματα, δηλαδή το γεγονός ότι ελέγχθηκε η κατάσταση ως προς τους εσωτερικά εκτοπισμένους και έτσι αντιμετωπίσαμε την κατάσταση υγείας και υγιεινής. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι επίκυνται ε, κυκλώνες. Ε, χιλιάδες... Ε, ε, Μουσαμάδες διανεμήθηκαν έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να αντισταθούν στις κακές καιρικές συνθήκες. Χιλιάδες τέντες διανεμήθηκαν έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν τους κυκλώνες. Οι πρόχειροι καταβλισμοί καθυστέρησαν, γι' αυτό καθυστέρησε και όλη η διαδικασία επειδή δεν υπάρχει και γη αυτή η επανακατανομή προσκρούει στην έλλειψη ε, γεών και γι' αυτό η Διασπορά χρειάστηκε να πάρει όλα τα αγροτεμάχια του νησιού. Επίσης τα χαλάσματα πρέπει να απομακρυνθούν, 20 εκατομμύρια κυβικά πρέπει να απομακρυνθούν, δηλαδή χρειάζονται 6 με 10 χρόνια με βάση τους παρόντες ε, ρυθμούς. Δεν έχουν παρά μικρά καροτσάκια και φαράσια οι κάτοικοι, άρα δεν μπορούν αυτά τα πενιχρά μέσα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες, χιλιάδες τόνους ε, χαλάσματα και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, να απομακρυνθούν με μικρές χειράμαξες. Η Ενδιάμεση Επιτροπή για την Ανοικοδόμηση της ΑΕΤΙΣ που έχει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό των περιορισμών τώρα έχει αρχίσει με τις εργασίες της και η εντολή αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων μόνο μερικά, μερικές εκατοντάδες ε, χιλιάδες δολάρια έχουν δοθεί σε σχέση με τα δέκα δις που είχαν υποσχεθεί οι δωρητές. Οι Αμερικανοί αναλαμβάνουν αυτό το έργο μέσω της ενδιάμεσης Επιτροπής Συντονισμού για την εκτέλεση του έργου, ενώ οι Ευρωπαίοι θέλουν μία ελαφριά δομή που να συνεργάζεται με τα Υπουργεία της ΑΕΤΙΣ. Αυτή η τελευταία προσέγγιση σημαίνει ότι συμμετέχουν τα Υπουργεία εξ αρχής, διότι η Επιτροπή έχει εντολή 18 μηνών. Θέλουμε να ενισχύσουμε μακροχρόνια την δυνατότητα συμμετοχής των Υπουργείων και να αλλάξει η μέθοδος εργασίας. Εμείς ως βασικός δωρητής θα πρέπει να έχουμε ηγετικό ρόλο. Επίσης εκφράσαμε την ανησυχία μας, διότι δεν υπάρχει ηγεσία και θα πρέπει να συμμετάσχουν, να συμμετάσχουν οι τοπικές αρχές στη διαδικασία νοικοδόμησης. Η διεθνής κοινότητα φαίνεται αισιόδοξη έναντι της δυνατότητας ε, μιας διαδικασίας εκλογών που προβλέπεται το Νοέμβριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ανέλαβαν μια κοινή προσέγγιση στον προγραμματισμό του 1,2 δις ε, ευρώ ε, από τη διάσκεψη της Νέας Υόρκης, 460, ε, από τα 460, 460 εκατομμύρια έχουν δοθεί μόνο 125 εκατομμύρια επί του παρόντος σε σχέση με την ενίσχυση των δυνατοτήτων ε, ανάκαμψης και ανοικοδόμησης. Η Επιτροπή αναθεωρεί αυτό το έγγραφο στρατηγικής μέχρι το τέλος του 2010 για την ανοικοδόμηση της IT και φαίνεται ότι οι αρχική τομείς υποδομής διακυβέρνησης δημοσιονομικής υποστήριξης αφορούν την ε, ε ανοικοδόμηση μετά το σεισμό και μέσα στα πλαίσια της διατροφικής ασφάλειας. Στις 2.30 στο, στην αίθουσα 1Ε1 θα έχουμε ένα γεύμα εργασίας με τους αντιπροσώπους της ΑΕΤ για την κατάσταση μετά το σεισμό και τη διατροφική ασφάλεια με εκπροσώπους από την ΑΕΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είσαστε ευπρόσδεκτοι στις 2.30 όπως σας είπα. Επίσης θα παρακολουθήσουμε την ε, ανθρωπιστική βοήθεια, όντας πολύ προσεκτική στην χρήση των πόρων και την αποτελεσματικότητα και τη διάφυγια του συστήματος που έχει τεθεί σε εφαρμογή. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στίφλερ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα μας ενημερώσατε για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός της Ε, Ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη δημοσιότητα ε, και κατά τα φαινόμενα τίποτα δεν πρόκειται να επιτευχθεί αν δεν γίνει μια μεγάλη φασαρία. Προτείνω λοιπόν να γράψουμε στον Bill Clinton και στον Πρωθυπουργό της Αιτής και να τους πούμε και να τους στείλουμε την έκθεσή μας με ένα συνοδευτικό γράμμα που θα προτείνουμε τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Ο κύριος Μπέρμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση Μισελ. Όταν συγκρίνουμε τα συμπεράσματά σας με το ψήφισμα το οποίο υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τον, ε, στις 10 Φεβρουαρίου, έχετε την εντύπωση ότι ουσιαστικά ελήφθη υπόψη αυτό το ψήφισμα συγκεκριμένα, δηλαδή ένα από τα βασικά θέματα στο ψήφισμα είναι η περίθαλψη των παιδιών και το πρόβλημα σχετικά με ε, τα ορφανά και την υιοθέτηση των ορφανών έχει ληφθεί κάποιο μέτρο για αυτά τα παιδιά. Το ψήφισμα αυτό ασχολείται με την εξασφάλιση ε, των καυσίμων για την κίνηση των φορτηγών των αυτοκινήτων. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτό το σημείο. Έχετε την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει αυτή την ηγεσία ή πιστεύετε ότι απλώς διατυπώνεται μία ευχή και ελπίζετε ότι θα υλοποιηθεί. Και τέλος, μιλάτε για τους τρόπους εκαθαρίσεως των ερηπείων. Ε, υπάρχουν ε, μόνο καροτσάκια. Μπορεί η Ευρώπη να κάνει μία επιπλέον προσπάθεια. Έχετε κάτι να μας υποδείξετε. Πριν απαντήσει η κυρία Στίφλερ, θα ζητήσω από ένα άλλο μέλος της αποστολής που πήγε στην Αϊτή, κύριε Τυρολιά. Ε, μήπως θέλετε κι εσείς να πείτε λίγα λόγια σχετικά με τις παρατηρήσεις σας. Απλώς θέλω να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως με όσα είπε η κυρία Στίφλερ. Η έκθεση ε, ήταν ε, πιστή σε αυτά τα οποία διαπιστώσαμε. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ λεπτή στην ΑΕΤ και θα μπορούσα να πω ότι είναι κρυκτική. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν πώς ίσως θα μπορούσε να ανάψει κάποια φωτιά από τη μια στιγμή στην άλλη και ε, δεν υπάρχει όπως είπε η κυρία Στίφλερ πολιτική ηγεσία. Είναι αληθές, το διαπιστώνουμε και έχουμε την εντύπωση άλλωστε ε, ε, έθεσα το ερώτημα στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και αντελήφθηκα ότι αυτές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις δικούν. Υπάρχει πλήρη έλλειψη κυβερνήσεως στην ΑΕΤ, δεν φαίνεται πουθενά και είμαστε μόνο λίγους μήνες από τις επικείμενες εκλογές. Το Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου προβλέπονται οι προεδρικές εκλογές στην ΑΕΤ αλλά παρόλα αυτά δεν βλέπουμε καθόλου τους πολιτικούς και εξεπλάγιν. Έπρεπε την Παρασκευή να τους ε, συναντήσουμε, να δούμε τους ε, διάφορους υπουργούς. Βέβαια είχαμε ένα πρόβλημα με τα αεροπλάνα, αλλά φαντάστηκα ότι την επομένη θα προσπαθούσαν να μας συναντήσουν και να συζητήσουν μαζί μας. Είδαμε και τον δήμαρχο του Πόρτο Πρανς, ε, τον είχαμε δεχθεί εδώ πριν από μερικές εβδομάδες αλλά επιτόπου δεν τον είδαμε καθόλου, δεν έχει έρθει σε επαφή με την αντιπροσωπεία μας και δεν έχει ε, χρησιμοποιήσει αυτές τις δυνατότητες μετακινήσεώς μας για να μας δείξει πώς είναι η πραγματικότητα. Είναι μια αποκεφαλισμένη κυβέρνηση και επίσης έχει πρόβλημα, ε, το, ε, έχουμε πρόβλημα με, τις, με το θέμα της γλώσσας, της επικοινωνίας. Έχουν εγκαταλείψει τα πάντα στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ιδίως το θέμα της ακίνητης ιδιοκτησίας το οποίο επισήμανε η κυρία Στίφλερ και εάν ε, καθαριστούν τα ερήπια δεν ξέρουν πού μπορούν να μπουν ε, όλα αυτά τα, τα θρήματα. Ε, επίσης την παραμονή των εκλογών δεν είναι σε θέση να λάβουν μία απόφαση ενώ είναι επίγον το θέμα. Ε, ανακοινώνεται η εποχή των κυκλώνων και νομίζω ότι είναι πολύ ανησυχητική η προοπτική, διότι όλα μπορούν να εκραγούν από τη μια στιγμή στην άλλη ή να διαταραχτούν. Είναι στην ΙΑΙΤ, είναι οι γειτονέ μου. Ξέρω ακριβώς τι γίνεται στη χώρα αυτή. Και όπως σας είπα, είναι σχετικά ήρεμη η κατάσταση. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν κάνει ε, σημαντική εργασία ακόμη και αν δεν είναι πολύ εμφανής. Αλλά προς το παρόν πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια επανάσταση στην ΑΕΤ. Μέχρι στιγμής έχουν τρόφιμα, αναλαμβάνεται η υγειονομική περίθαλψη, δεν υπάρχει επιδημία, είναι σε επαφή με μονάδες υγειονομικής, υπάρχουν επιτόπου γιατροί, ε, δηλαδή στο κάτω-κάτω της γραφής μέχρι στιγμής δεν κινούνται οι αιτινοί. Φοβόμαστε όμως ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου και όλα αυτά μπορούν να συμβούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Όσον αφορά την ανοικοδόμηση, όπως αναφέρθηκε, είναι το πιο δύσκολο, το πιο σοβαρό θέμα και πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασκήσει όλες τις δυνατές πιέσεις ώστε να υλοποιηθεί και να κινητοποιηθεί αυτή η επιτροπή, η προσωρινή επιτροπή για την ανοικοδόμηση της ΑΙΤΙΣ. Τα έγγραφα τα οποία παρουσίασε η κυβέρνηση της ΑΙΤΙΣ ε, δεν είναι όντως ε, λειτουργικά και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε με κάθε τρόπο και ε, όντως ανησυχούν μεταξύ ε, της αμερικανικής λύσεως και ε, της ευρωπαϊκής λύσεως. Δηλαδή ε, για την αμερικανική λύση μία προσωρινή επιτροπή η οποία όμως αποκλεί ουσιαστικά τους αιτινούς και την ευρωπαϊκή λύση η οποία είναι πιο περιορισμένη ίσως αλλά η οποία θα επέτρεπε στους αιτινούς να συνεργαστούν με ε, αυτούς οι οποίοι τους διαθέτουν τους χρηματικούς πόρους και θα επιτρέψει στους αιτινούς να αναλάβουν τη σκητάλη διότι η εντολή είναι 18 μηνών. Υπάρχει λοιπόν ο δισταγμός αυτός μεταξύ των δύο συστημάτων, δεν μπορώ εγώ να σας πω, ε, δηλαδή ε, δεν ξέρω πώς οι αιτινοί θα μπορούσαν να δουλέψουν καλύτερα με τους άλλους δανειοδότες του και να αναλάβουν τη σκητάλη στη συνέχεια. Πιστεύω όμως ότι είναι ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να συζητείται και πρέπει να δούμε. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επέμβει δραστήρια για να μπορέσει να υπάρχει επιτάχυνση. Επίσης η κατάσταση της ΑΙΤΙΣ είναι πολύ περίπλοκη διότι η πόλη του Πόρτο Πράνς επλήγει ε, πολύ άσχημα, ε, έχει μεγάλες δυσκολίες από πλευράς τοπογραφικής της πόλεως και θα έπρεπε να μπορέσουμε τουλάχιστον στον τομέα αυτό να μαζέψουμε όλα τα χαλάσματα, να καθαρίσουμε το Πόρτο Πράνς γιατί δεν είπαμε ότι το Πόρτο Πράνς είναι απίστευτα βρώμικο, δεν υπάρχει καμία συνειδητοποίηση ότι χρειάζεται ένα περιβάλλον το οποίο να είναι υγιεινό. Γίνεται οτιδήποτε εκεί, δεν υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει πλήρης αναρχία. Το μόνο το οποίο είναι θετικό σε όλα αυτά είναι ότι η ζωή ε, έχει ξαναξεκινήσει, έχει πάρει το δρόμο της και βλέπουμε πράγματι ε, ότι υπάρχουν ε, μικρά εμπόρια ε, και δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό το δράμα διότι μπροστά στο, στο προεδρικό μέγαρο υπάρχουν τουλάχιστον 10.000 άτομα σε τέντες. Η κατάσταση λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολη, θα πρέπει να παρέμβουμε, κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να ε, αλλάξουμε τον ρου των πραγμάτων. Ε, όσον αφορά την ενέργεια θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των αιτινών και αυτό είναι πήγον διότι αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να αποψηλώνουν τα ε, δάση και ε, ε, διότι χρειάζονται ξύλα οπότε είδαμε μπροστά σε όλα τα αρτοπία ότι υπάρχουν βουναλάκια ε, ξύλο, ξυλίας για να μπορέσουν να έχουν κάποια ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να επιληθεί τουλάχιστον αυτό το πολύ βασικό θέμα και να μπορέσει η κατάσταση να εξελιχθεί θετικά, διαφορετικά θα υπάρξει μια καταστροφή. Οι κυκλώνες, οι εκλογές είναι δύο πιτιδαποθήκες οι οποίες θα, θα πρέπει να κατασταλούν το πιο γρήγορα δυνατόν. Ευχαριστώ κύριε Τυρολιά. Αυτό είναι τρομακτικό. Η κατάσταση αυτή είναι τρομακτική. Και τώρα αρχίζω να αντιλαμβάνομαι, διότι εδώ μεν τραβάμε τα μαλλιά μας και είδα το ίδιο με το τσουνάμι και ε, ε, θέλαμε να παρακολουθήσουμε την πορεία του τσουνάμι και μετά από δύο ε, χρόνια στην Ινδονησία και στην Σρι Λάνκα ξεκίνησε η κατάσταση να κινείται. Αλλά ε, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες πηγαίνουν εκεί, ανθρωπιστές, ε, επισκέπτονται και μετά από δύο-τρεις εβδομάδες όλοι έχουν εγκαταλείψει το σοβαρό πρόβλημα ε, που είναι ότι χρειάζεται βιώσιμη εξέλιξη χρειάζονται μπουλντόζες παραδείγματο χάρη. Ε, δεν είναι δυνατό να μεταφέρει κανείς όλα αυτά τα χαλάσματα με τα χέρια, αλλά ο κύριος Κλίντον είναι ο συντονιστής. Οπότε εγώ διατυπώνω μία πρόταση. Κυρία Στίφλερ, εσείς βέβαια ε, δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε ή θα ρωτήσω άλλους να παλάμουν το λόγο πριν από σας. Θέλετε να κάνετε μία συνέντευξη τύπου της Επιτροπής και να κάνετε μεγάλη φασαρία ε, για αυτή την ε, έλλειψη ενημερώσεως των μέσων και να χρησιμοποιήσετε την Επιτροπή μας ε, για να κινητοποιήσετε την κατάσταση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήγαν στην ΑΙΤ με την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Ήταν εξαιρετική η έκθεση που συνέταξαν, ε, όπως διαπίστωσα τώρα. Θυμάμαι όταν κάναμε την πρώτη συζήτηση για την ΑΕΤ εδώ, είχα τονίσει πως πραγματικά πρόκειται για μεγάλη καταστροφή, για φλέγον θέμα, αλλά καθημερινά υπάρχουν τέτοιες καταστροφές ανά τον κόσμο, σε διάφορα μέρη του κόσμου όταν προσπαθούμε να διαπιστώσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί, οφείλουμε να κάνουμε και ρεαλιστικές αξιολογήσεις. Εξ αρχής λοιπόν, αυτό πίστευα, ίσως είναι υπέρμετρες οι φιλοδοξίες μας. Είναι αδύνατον ε, να νοικοδομήσουμε μια κατεστραμμένη χώρα εκ του μειόντος. Πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές και να δούμε ποια μπορεί να είναι η επίπτωση της ε, βοήθειας, της συνδρομής της Ένωσης. Συμφωνώ με τον Μπέρναντ Πρέπει να ιεραρχήσουμε συγγνώμη, τις προτεραιότητές μας. Δηλαδή, σε ποιους τομείς πρέπει να εστιάσουμε τη συνδρομή, την παρέμβασή μας για να είμαστε αποτελεσματικοί. Σαφέστατα δεν θα είμαστε όλοι αποτελεσματικοί. Υπάρχουν ε, διασκέψεις, ε, υψηλά κλιμάκια που έχουν μεταβεί ήδη στην ΑΕΤ, αλλά δεν έχουν ε, σημειώσει αποτελεσματική δράση. Η είναι ένα ανήμπορο, φτωχότατο κράτος εγκαταλελειμμένο από τις ε, γειτονικές χώρες ε, που ε, είτε πρόκειται για ισχυρές είτε για αδύναμες γειτονικές χώρες. Είναι μια φυσική αδικία σε εισαγωγικά να πλήτεται η πλέον φτωχή χώρα από αυτή την καταστροφή. του λεχθέντος πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, ξαναλέω να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας. Όπως είπε και ο συνάδελφος Μπέρμαν, υπάρχει αυτό το θέμα των χαλασμάτων και των φορτηγών Ορίστε, να ένα σημείο όπου μπορούμε να έχουμε απτά αποτελέσματα, να είμαστε αποτελεσματικοί. Ας μην προσπαθούμε να ε, τροφοδοτούμε αυτή την ε, φιλοδοξία μας, ε, δηλαδή νυχθημερό να νοικοδομήσουμε τη χώρα. Είναι ανέφικτο αυτό, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Ας παραμείνουμε γαλήνοι και να προσπαθήσουμε να έχουμε αποτελεσματική δράση σε όποιο τομέα και αν παρέμβουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ήταν σοφά τα λόγια σας. Well, I've listened, Ο κύριος Νιούτον Ντάν. Ε, είμαι αποτροπιασμένος. Ε, φυσικά επίκειται καταστροφή με τους κυκλώνες, ε, τις βροχές κτλ. Ο Μπιλ Κλίντον είναι υπεύθυνο, τουλάχιστον κατ' όνομα. Γιατί δεν τον καλούμε στην Επιτροπή για να μας απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Εμείς δίνουμε τα κονδύλια, αλλά τι τα κάνει τα κονδύλια. Σε έρθει να μας εξηγήσει. Anybody else to make a contribution before I ask the Commission to make their contribution. Θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά την κυρία Στίφλε που θα κάνει τις ε, καταληκτικές παρατηρήσεις εκτός και αν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που επιθυμούν να παρέμβουν στη συζήτηση. Who in the commission? Christoph Gadry. Ο Κριστόφ Γκάντρι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Μαριάν Λεμόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την αναφορά της αντιπροσωπείας μετέβη στην ΑΕΤ. Θα θυμάστε ίσως ότι στη διάσκεψη των δωρητών η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για ένα ποσό άνω των 2,2 δις ε, και η Επιτροπή είχε υποσχεθεί 460 εκατομμύρια. Τι συνέβη λοιπόν σε αυτούς τους 6 μήνες πάνω από 300 εκατομμύρια από 460 έχουν ήδη δρομολογηθεί από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις εβδομάδες που ακολούθησαν το σεισμό, Έχουμε ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων ε, για να αποκαταστήσουμε τις ε, ικανότητες ε, της λειτουργίας του κράτους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο ώστε η κυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα να δράσει και να αναλάβει την ηγεσία της διαδικασίας ανοικοδόμησης. 35 εκατομμύρια σε άμεση δημοσιονομική στήριξη έχουν ήδη εκταμιευθεί ε, στο τομέα της υγείας και για να καλυφθούν οι πλέον επίγουσες δαπάνες ε, μετά την καταστροφή. Ε, υπάρχει όμως ένα δημοσιονομικό κενό ακόμη στην ΑΕΤ, στον προϋπολογισμό της ΑΕΤ, οπότε για το 2010 έχουμε προβλέψει και άλλες πληρωμές. Επίσης αρχίσαμε την ανοικοδόμηση πέντε υπουργείων που καταστράφηκαν 90% καταστράφηκαν ε, στον σεισμό, αλλά εμείς έχουμε αρχίσει την ανοικοδόμηση των πέντε βασικών υπουργείων για τα δημόσια έργα, για την παιδεία, το Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Εμπορίου και Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων. Επίσης, ε, έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα για να συνδράμουμε την κυβέρνηση της ΑΕΤ ε, ούτως ώστε να μπορεί να δράσει και να αντιμετωπίζει τις κρίσεις όταν συμβαίνουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στο, στην περίοδο των κυκλώνων γιατί όλοι μένουν σε αυτοσχέδιους καταβλισμού, σε αντίσκηνα και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δυνατότητα της κυβέρνησης ε, ε, να κατοχυρώσει την πολιτική προστασία. Ε, και φυσικά αυτό αφορά και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Επίσης χορηγούμε κονδύλια μέσω του ΟΗΕ ε, για το πρόγραμμα Cash for Work, μετρητά για εργασία, δηλαδή για να ε, μην παραμένουν βαθείς οι πληθυσμιακές ομάδες να μπορούν να έχουν κάποιες αποδοχές. Για τα υπόλοιπα τώρα εκατομμύρια που, για τα οποία έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έχουμε υπογράψει πέντε χρηματοδοτικές συμφωνίες ε, όταν ο Αρμόδιος Επίτροπος μετέβη τον Απρίλιο στην ΑΕΤ. Τα προγράμματα αυτά σχετίζονται με τις υποδομές, οδικό δίκτυο, υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, χωροταξική ανάπτυξη και δημοσιονομική στήριξη ε, συνεχίζουμε να υλοποιούμε τα προγράμματα στην ΑΕΤ και συζητούμε με τις αρχές ε, ούτως ώστε να επαπαπροσανατολίσουμε κάποια διαθέσιμα κονδύλια ούτως ώστε ε, να ε, προσαρμοστούν καλύτερα στο σενάριο, στο πρόγραμμα νοικοδόμησης. Τα υπολοιπόμενα κονδύλια από τα 460 εκατομμύρια προγραμματίζονται τώρα σε μια κοινή άσκηση που ε, με τις αρχές της ΑΕΤ και τα κράτη-μέλη ε, θα έχουμε λοιπόν ένα νέο ε, έγγραφο στρατηγικής και ένα νέο πρόγραμμα δράσης και έτσι η κοινωνία των πολιτών και η κυβέρνηση της ΑΕΤΗΣ ε, θα συμμετάσχουν στην διαδικασία προγραμματισμού και θα αρχίσουν να τρέχουν τα νέα προγράμματα από το φθινόπωρο το 2010. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν πάρα πολύ ακριβής και λίγα ενημερωτική η παρουσίασή σας. Νομίζω ότι πρέπει να τα σημειώσουμε όλα αυτά ε, σε μια επιστολή προς τον ε, ε, πρόεδρο Κλίντον για να γνωρίζουμε πώς ακριβώς χρησιμοποιεί τα κονδύλια της Ένωσης. Η κυρία Στίφλερ. Θέλει κάποιος άλλος να κάνει ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή έχουμε χρόνο, μήπως έχετε άλλες ερωτήσεις. Merci Κυρία Στίφλε, για να απαντήσω στον κύριο Μπέρμαν ε, για την περίθαλψη των παιδιών. Ε, επισκεφτήκαμε ορφανοτροφία όπου υπάρχουν ε, ε, παιδιά που είναι πραγματικά ορφανά και παιδιά που έχουν ακόμη τους γονείς τους, οι οποίοι όμως δεν μπορούν πλέον να τα φροντίσουν, να τα μεγαλώσουν, να τα αναθρέψουν. Ε, είναι τυχερά τα παιδιά που είναι στα ορφανοτροφία γιατί μπορούν να φάνε, ε, έχουν ρούχα, ε, έχουν που να κοιμηθούν. Το βασικό πρόβλημα είναι οι υιοθεσίες έχουν παρεμποδιστεί οι αιτήσει για υιοθεσία πριν το σεισμό γιατί θα έχετε ακούσει ότι υπήρξαν ε, απαγωγές ε, παιδιών ε, δεν υπάρχουν τα μέσα για να χειριστούμε διαφορετικά τα αιτήματα πριν και μετά το σεισμό. Ο πρέσβης της Γαλλίας, ο πρέσβης στη Γαλλία με διαβεβαίωσε ότι μέσα σε 8 ημέρες θα συνεχιστεί η διαδικασία και θα αρχίσουν να γίνονται υιοθεσίε. Τα παιδιά ε, που μένουν ε, στα αντίσκηνα, στο Πόχο Prince ε, ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Υπάρχει τώρα ένα σύστημα που έχουν φτιάξει οι γονείς και ονομάζεται αυτό το πρόγραμμα «Μένουν μαζί τα παιδιά». Τι σημαίνει αυτό, ότι τα παιδιά μένουν σε ένα αντίσκηνο ε, και πηγαίνουν στον Άγιο Δομήνικο παραδείγματος χάρη όπου υπάρχει ε, εκμετάλλευση των ε, παιδιών πρόκειται για δουλεία και είναι ένα φλέγον πρόβλημα, επίκαιρο δυστυχώς. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν βάλει τα δυνατά τους, αλλά η κατάσταση έτσι έχει, γιατί οι γονείς δεν μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά τους, οπότε τα δανείζουν σε εισαγωγικά προσωρινά μέχρι να βρουν τα προστοζήν. Ε, ε, για τα παιδιά λοιπόν έτσι έχει η κατάσταση. Ε, για τα καύσιμα δεν υπάρχουν. Είναι απλό. λίγα υπάρχουν, αλλά όχι πολύ περισσότερα σε σχέση με το παρελθόν. Το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτως ή άλλω. υπάρχουν μποτιλιαρίσματα τριών ωρών για να κάνει κανείς ένα ή δύο χιλιόμετρα. είναι αδύνατο σχεδόν να μετακινηθεί κάποιο στο Πόγο Πχάνσε. Ε, τώρα, αν έχει αναλάβει την ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα ότι κάνει ό,τι μπορεί η Ένωση. Συναντηθήκαμε με ε, υπαλλήλου Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εργάζονται σε απίστευτε συνθήκε. Ε, οι υπάλληλοι των μη κυβερνητικών οργανώσεων έχουν ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό το προσωπικό του ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειώσει το προσωπικό της, ε, η Ευρωπαϊκή Μητροπή λειτουργεί μέσα σε ένα σπίτι που τους έχει δανείσει η κυβέρνηση. Φυσικά δεν υπάρχει διασύνδεση με το διαδίκτυο, δεν υπάρχει κλιματιστικό, δεν υπάρχει τίποτα ε, είναι αδύνατον να ε, δουλέψει κανείς αυτές τις συνθήκες. τώρα με ρωτήσατε αν έχει ηγετικό ρόλο η Ένωση. Κάνει ό,τι μπορεί, σας ξαναλέω. Ε, πρέπει όντως ε, να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους στην ΑΕΤ, αλλά είναι σε τέτοια κατάσταση η χώρα που είτε μιλάμε για την Ένωση, είτε μιλάμε για τη ΣΥΠΑ, κάποιος πρέπει να κινηθεί, δεν γίνεται να συνεχιστεί έτσι, ε, να παραμείνει έτσι η κατάσταση για την ανοικοδόμηση θα έλεγα ότι οι θύνοντες και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε την κοινή λογική ορισμένες φορές. Η κυρία Μαριέλ, δεν ξέρω πώς ε, είναι το επίθετό σας, συγγνώμη, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας μιλούσε για την ανοικοδόμηση και μας είπε ότι υπάρχουν σχέδια ε, αποκατάστασης των υποδομών, αποκατάστασης του δικού δικτύου κτλ. Μάλιστα, θα έλεγα ότι το πλεονέκτημα που έχει ένα τσουνάμι σε σχέση με αυτό το σεισμό είναι ότι το τσουνάμι τα πήρε και τα σήκωσε όλα. Ε, ε δεν γίνεται τώρα όμως που υπάρχουν τα χαλάσματα να ανοικοδομήσουμε το οδικό δίκτυο. Ε, με τον σεισμό, είτε μιλάμε για την Ένωση, είτε μιλάμε για τη ΣΥΠΑ, ε, πρέ, χρειάζονται οι μπουλντόζες, ε, πήγαν οι μπουλντόζες για να βγάλουν τα... Ε, ε, πτώματα για να βγάλουν τους πολίτες από τα χαλάσματα και τελικά τι έγινε, έφυγαν οι μπουλντόζες μετά είναι ό,τι πιο ηλίθιο, συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι, μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί και πώς έγινε αυτό. Εκατομμύρια ευρώ δαπανίσαμε και να πάνε τα μηχανήματα εκεί πέρα και μετά τα ξαναφέραμε στις χώρες μας στο World Trade Center στη ΣΥΠΑ δύο χρόνια χρειάστηκαν για να βγάλουν τα χαλάσματα και μιλάμε για τη ΣΥΠΑ. Φανταστείτε πώ τόνους ερήπια ε, έχουμε στο πόρο πράνση και τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε τα καροτσάκια και τα φτιαράκια και προσπαθούμε να τα βγάλουμε. Μα είναι αδύνατον. Έχουμε φύγει όλοι και πήραμε μαζί τις μπουλντόζες μας ε τα φορτηγά μα. Σήμερα λοιπόν είναι αδύνατον να καταρτήσουμε σχέδια δράσης στο μέτρο που εξακολουθούν να υπάρχουν τα χαλάσματα. Έλεγε ο κύριο Τυρολιά ότι αρχίζουν τα μικρά μαγαζιά να ξαναλειτουργούν. Τα μαγαζιά ξέρετε ότι ε, ε, φτιάχνονται πάνω στα χαλάσματα, μα είναι αδιανόητο αυτό που βλέπει κανεί ε, στο Πόρτο Πράνσε. Και αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, και συμφωνώ με τον κύριο Βερέτ, θα πρέπει με τα χρήματα που έχουμε συλλέξει να ξαναφέρουμε τις μπουλντόζες, να ξαναφέρουμε τα φορτηγά του, ε, τους μηχανικούς, ε, τους εργολάβους. Δεν μπορούν οι άνθρωποι στην ΑΕΤ να κάνουν ε, κάτι δομημένο και η κατάσταση ήταν καταστροφική και πριν γιατί δεν μπορούν. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Είναι, συγγνώμη, είναι λυπηρό, αλλά ας το παραδεχτούμε για να προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε φορτηγά, ε, μπουλντόζες, εργολάβους, εργάτες που ξέρουν να λειτουργήσουν ένα εργοτάξιο. Ε, αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Τώρα θα, σε σχέση ένα λεπτάκι να δω αυτά τα είπα. Υπάρχει και κάτι καλό, το Cash for Work, αυτό το πρόγραμμα μετρητά για εργασία. Ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει τον δρομολόγησαν, 100 ε, δολάρια την ημέρα παίρνουν οι Αιτιανοί για να δουλέψουν για την ανοικοδόμηση. Σας διαβεβαιώ ότι 20 χρόνια θα χρειαστούν να συνεχίσουμε έτσι. Λοιπόν, για τις ε, συνεντεύξεις τύπου, το αντίθετο, εγώ πιστεύω, πρέπει να παρενοχλήσουμε τον τύπο να προκαλέσουμε τον τύπο. Δεν είναι φυσιολογικό που, σταματήσαμε να μιλάμε για την ΑΕΤ. Κανεί δεν ασχολείται τώρα με την ΑΕΤ. Όταν γύρισε, έστειλα ανακοινοθέντα τύπου στον τοπικό τύπο. κανένα δεν τα δημοσίευσε, Κανεί δεν ενδιαφέρεται. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω κάτι παραπάνω. Ε, να πω κάτι παραπάνω. Ο τύπος ε, είναι υπεύθυνο γιατί ενδιαφέρεται μόνο για κάτι πιο ε, ανάλαφρο που ίσως ε, που λέει περισσότερε εφημερίδε. Εμεί πρέπει να προκαλέσουμε τον τύπο γιατί ο τύπο αποφασίζει τι θα κάνουμε για τέτοιες χώρες. Εγώ ε, ε, προτίθεμαι να παρενοχλήσω τον τύπο. Για τον κύριο Κλίντον το έχω προβλέψει ήδη και θα σας το πρότεινα να ε, στείλουμε μια επιστολή στον κύριο Κλίντον που είναι ε, επικεφαλής ε, της ενδιάμεσης επιτροπής ε, που είναι ε, αποτελεσματική σε ανησυχητικό, αναποτελεσματική σε ανησυχητικό σημείο. Για να γίνω και πιο κακιά θα έλεγα ότι δεν, δεν τα καταφέρνουν. Ε, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης ενδιαφέρονται μόνο για τις τοπικές εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο, τα υπόλοιπα, ε, αυτοί που είναι στα αντίσκηνα είναι μέρος, ε, τι να σας πω, του τοπίου στο Πόγο Πχάνς, κανείς δεν ασχολείται. Ο πρέσβης στο Πόγο Πχάνς, ωραία, συμπαθητικός είναι, αλλά ξέρετε, μίλαγε λέγοντας, εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η IT, δεν είναι ότι απλώς σηκώνουν τα χέρια ψηλά, μυρολατρούν σε απίστευτο σημείο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να πιέσουμε, να στείλουμε επιστολή ε, στον πρόεδρο Κλίντον, Ακόμη και έτσι, μάλλον δεν τα καταφέρουμε. Κινδυνεύουν τα παιδιά. Εάν δεν κάνουμε εμεί κάτι, τίποτα δεν θα γίνει. Ζητώ λοιπόν ε, να χρησιμοποιήσουμε την κοινή λογική, να φέρουμε τα μηχανήματα, να φέρουμε του εργάτε και μόνο μετά ε, μπορούμε να αρχίσουμε να ε, φιλοσοφούμε για την ανοικοδόμηση. Πριν απομακρυνθούν τα χαλάσματα, δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για ανοικοδόμηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε και την κυρία Στίφλερ για τα πολύ στεναρά της λόγια. Θα ήθελα η Επιτροπή να μας απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα που απασχολεί όλους τους συναδέλφους σε αυτή την αίθουσα. Γιατί ε, αυτά τα, τα bulldozer απομακρύνθηκαν χωρίς να συμπληρώσουν, να αποπερατώσουν το έργο τους. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτή τη δύσκολη ερώτηση. Οι περισσότερες μπουλντόζες ανήκαν στις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μας. Ε, οι ένοπλες δυνάμεις εγκατέλειψαν τη χώρα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο απομακρύθηκαν και οι μπουλντόζες γιατί αποτελούν τμήμα του στρατιωτικού σκέλους των κρατών. Αυτό όμως δεν μας διδάσκει κάτι για το μέλλον, λέει ο πρόεδρος. Δηλαδή από τη μία πλευρά λέμε, η κοινωνία των πολιτών αντιδρά όταν επεμβαίνουν οι στρατιωτικές δυνάμεις. Απ' την άλλη φορά όμως χρειαζόμαστε αυτά τα μέσα γιατί πολλές φορές λέμε ότι ε, χρειάζονται ε, μεγάλα μέσα για να απομακρύνουν αυτά τα χαλάσματα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό χωρίς αυτή τη, την υποδομή. Δεν νομίζω ότι οι στρατιωτικοί εγκατέλειψαν την ΑΕΤ γιατί η κοινωνία των πολιτών αντέδρασε. Τα πράγματα λειτουργήσαν καλά. Ήταν πολιτική απόφαση και απόφαση του, των ενόπλων δυνάμεων και δεν ελήφθη μετά από πιέσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων ή της κοινωνίας των πολιτών. Ήταν και οικονομική η απόφαση, οικονομικής φύσης. Ποιος έλαβε την απόφαση. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση οι αποφάσεις ελήφθησαν από τον πρόεδρο Ομπάμα, ο οποίος απομάκρυνε τις στρατιωτικές δυνάμεις πρόσφατα. Πρέπει να ρωτήσετε τα κράτη-μέλη γιατί οι στρατιωτικές δυνάμεις που ήταν υπεύθυνε για την απομάκρυνση των χαλασμάτων απομακρύνθηκαν. Τι ρωτάτε εμένα. Θα ήθελα να γίνει ε, δεύτερος γύρος συζητήσεων, αν κάποιος θέλει να λάβει το λόγο. So, uh, Mrs. Stifler, thank you for... Στη κυρία Στίφλερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετική εισήγηση. Θα πρέπει όμως να κάνουμε περισσότερα, να υπάρξει συγκεκριμένη δράση και ε, ακούσαμε και τις συστάσεις της κυρίας Στίφλερ και να υποβάλουμε και ερωτήσεις προς τα κράτη-μέλη που συμμετείχαν με μπουλντόζες, με ελικόπτερα, να ρωτήσουμε και την κυβέρνηση των ΙΠΑ και να τους πούμε, να τους ρωτήσουμε περί τίνος πρόκειται. Και ίσως να μπορέσουμε να αποστείλουμε μία ανοιχτή επιστολή για να οργανώσουμε και μία συνέντευξη τύπου για να επανέλθουν ε, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς επιτόπου. Ευχαριστώ. Μου ελέγχθη ότι μπορούμε να φύγουμε για το μεσημεριανό μας βγεύμα και θα είμαστε πίσω στις τρεις. Στις 3 διότι έχουμε τον κύριο Πίμπαλξ ο οποίος θα έρθει εδώ. στις 3 λοιπόν με τον κύριο Πίμπαλξ.